τη χρήση του χρόνου γιατί έχουμε και άλλα σημεία που θα μας απασχολήσουν πριν από το τέλος των εργασιών μας. που προβλέπεται μέχρι τις 6.30 θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα έγγραφο, ένα φάκελο που σχετίζεται με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων δυνάμει του κανονισμού του άρθρου 50. Και θα ήθελα να σας ε, ανακοινώσω ότι στις 10 Ιανουαρίου λίγη προθεσμία υποβολής τροπολογιών στις 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία από την Επίτροπή μας θα γίνει στις 3 Φεβρουαρίου του 2011. Δίνω λοιπόν το λόγο στην κυρία Γιαρόκα χωρίς άλλη καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα μετά τις πρώτες συζητήσεις όπως προβλέφθηκαν και με τις ε, άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές, την ε, ΚΑΛΤ και της απασχόλησης. Μιλάμε για, τις, ε, για την επένδυση στην εκπαίδευση των Ρωμά. Και επίσης το Κοινοβούλιο τόνισε και το θέμα της κατάρτισης και εκπαίδευσης, όπως ανέφερε και ο κύριος Πάκουλα. Όπως είπε και η κυρία Γκέν στην Επιτροπή Απασχόλησης, είχαμε μία πολύ καλή συζήτηση και το πρόγραμμα σύγχρηματοδότησης που προβλέπεται στη δική της γνωμοδότηση συνάδει με το δικό μου. Χαίρομαι διότι αυτές οι γνωμοδοτήσεις εντάσσονται στην έκθεση. Όπως είπε και ο κύριος Κόβατσεκ, στην τροπολογία που υπέβαλε και τη στιγμή που θα μιλήσουμε για τις απομακρυσμένες περιφέρειες, και του χρόνου. Ε, διανύουμε μια πολύ ε, κρίσιμη στιγμή έως ότου ε, εγκρίνουμε αυτή την στρατηγική. Η μελέτη που έχουμε αναθέσει στο College of London θα είναι έτοιμη την επόμενη Τετάρτη και θα ήταν σκόπιμο να βασίσουμε τις ε, τροπολογίες μας σε αυτή τη μελέτη. Από το έγγραφο εργασίας και μετά τα πιο σημαντικά έξι σημεία που θα ήθελα να θίξω αφορούν το, την αιτιολογική σκέψη του κειμένου θα πρέπει να έχουμε μια εσωτερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 που να αποτελεί συνδετικό κρίκο και να μην κάνει διαχωρισμούς. Ένα δεύτερο θέμα είναι τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή τη διαδικασία και όπως σας είπα πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εποπτεύει και να ελέγχει τη διαδικασία και από την ε, σύσταση αυτού του νέου σώματος δεν νομίζω ότι χρειάζεται να γίνει τίποτα επιπρόσθετο. Η παρούσα επιτροπή, ε, η προσωρινή επιτροπή εργασίας υπέν των Ρωμά θα πρέπει να μετατραπεί σε ένα μόνιμο σώμα. Επίσης μιλάμε για μια ετήσια έκθεση αξιολόγησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποβολή προτάσεων στο Συμβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και ένα βαθμολόγιο το οποίο θα πρέπει να ισχύσει. Το τέταρτο σημείο είναι ότι οι χώρες θα πρέπει να έχουν ένα διοικητικό σώμα ή έναν σύνδεσμο έναν εθνικό σύνδεσμο για να δούμε πώς μπορεί η ελεγκτική αρχή της Επιτροπής να δράσει άμεσα. Τώρα, από πού θα γίνει η χρηματοδότηση. Μέσα στα πλαίσια των Ταμείων Συνοχής θα μπορέσαμε να βάλουμε κατά μέρος, δηλαδή να έχουμε ένα προσυπόμνηση ή ένα αποθεματικό και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μεγιστοποιήσουμε τη χρήση των κονδυλίων για να υπάρχει άμεση διασύνδεση μεταξύ κατανομής και χρηματοδότησης. Γιατί θα πρέπει οι χώρες που ε, τα καταφέρνουν καλύτερα να λαμβάνουν και περισσότερα χρήματα. Δηλαδή να βασιζόμαστε στα αποτελέσματα για τη χρηματοδότηση. Και ως χώρες που θα ήθελαν να συμμετάσχουν, πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε και τις βαλκανικές χώρες που έχουν ε, ένα μείζον πρόβλημα σε σχέση με τους Ρωμά. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι γίνεται μετά το 90. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, αναλάβουμε το, θέμα από, από, την, από τις απαρχές του και μετά και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις βαλκανικές χώρες που αντιμετωπίζουν ένα παρόμοιο ζήτημα. Αυτά είναι τα σημεία που θεωρώ ότι είναι ύψης της σημασίας και θα πρέπει να μας απασχολήσουν γιατί αυτό είναι το πλαίσιο εργασίας που θα μας απασχολήσει για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις διακρίσεις και τη φτώχεια που υφίσταται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Γιαρόκα, εκτιμούμε ιδιαίτερα την εργασία σας. Τώρα ε, ξεκινούν οι συζητήσεις. Κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εργασία που έχει επιτελέσει. Αχρητούδε και υποστηρίζω πλήρω τα όσα είπε τώρα και τη δράση πρέπει να αναλυφθεί στη βάση της εκθεσεώς της. Πράγματι τώρα πρέπει να συνεργαστούμε και να δώσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα που η Επίτροπος Ρέντινγκ ανακοίνωσε το τι προτίθεται να πράξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα δεν μιλούμε πλέον από ό,τι φαίνεται για στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη των Ρώμα, αλλά για ένα πλαίσιο εθνικών στρατηγικών. Τι ωραία. 27 εθνικές στρατηγικές για, τον, ε, για τους Ρώμα, μα θα προκαλέσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή σύγχυση και αν μπορούσε κάποιο να δει τι θα γίνει μετά από 20 χρόνια, είμαι βεβαία ότι θα δει την ίδια ακριβώ κατάσταση. Άρα, είναι καιρό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για το, το πού βρισκόμαστε και το τι θέλουμε. Και όχι μοναχά μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά το ίδιο μήνυμα έχουν στείλει και όλες οι διασκέψεις κορυφής των Ρώμα εν προκειμένου και ανεξαρτήτως του, γεγονός ότι, του γεγονότος συγγνώμη, ότι εγώ θα υποβάλω κάποιες τροπολογίες, συμφωνώ απόλυτα με την θέση της συγγητρίας, όπως την εξέφρασε σήμερα. Ίσως την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο, όπου θα βρεθούμε με την Επίτροπο Ρέντινγκ, να έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε ορισμένες ερωτήσεις σε σχέση με αυτή την ιδέα του πλαισίου, διότι ε, νομίζω εκκρεμούν πολλές ερωτήσεις που ακόμη από εκείνο το όνειρο της Λίβια να υπάρξει δηλαδή μια νομική βάση για μια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα κατευθυνόμαστε προς κάποιο πλαίσιο κάποιων ασαφών πραγμάτων για το μέλλον. Νομίζω ότι πρέπει να δουλέψουμε επικοδομητικά όλοι προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και την εισηγήτρια σε μια πρώτη συζήτηση, σε ένα πρώτο γύρο συζητήσεως, είχαμε εκφράσει πολλές κριτικές. Είχαμε γίνει, είχαμε γίνει φτερά και πούπουλα, όπως λέμε. Θα έλθω όμως και στις λεπτομέρειες, αλλά υπενθυμίζω την πτυχή ανάμεσα σε μια εθνική καταγωγή, ρατσισμό και συγκεκριμένες διακρίσεις που είναι σημαντικά για τα όσα θα συζητήσουμε ακόμη. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τη διασύνδεση αυτή και κυρίως η θυμίζω και την παρέμβαση του Βαλέριο που και στην ακρόαση είχε καταστήσει σαφές ότι μπορούμε να αποφασίσουμε ό,τι θέλουμε και στον κοινωνικό και στον οικονομικό τομέα εάν όμως δεν αναγάγουμε σε αξία τον αντιτσιγκανισμό, την καταδίκη δηλαδή, του αντιτσικανισμού δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Επίσης, η κατάσταση των ανήλικων Ρωμά στις διάφορες ε, φάσεις της ζωής. Εδώ ίσως μπορούμε να αναπτύξουμε κάποιες νέες παραγράφους που να περιλάβουμε τα θέματα αυτά. Κάτι που για μένα είναι πολύ σημαντικό και είναι και το κυριότερο μήνυμά μου τώρα πώς θα καταφέρουμε ώστε οι χώρε μέλη να αναλάβουν περισσότερο τις ευθύνες τους. Όσο θαυμάσια και αν είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αναπτύξουμε, αν δεν καταφέρουμε να αυτοδεσμευτούν οι χώρε μέλη, να μην έχουν τη δυνατότητα δηλαδή με κάποιο τρόπο να διαφύγουν από την ανάληψη των ευθυνών τους, Αυτό έχει συζητηθεί και στην ακρόαση. Δηλαδή, εν τέλει, τα πράγματα που θα συμβούν θα συμβούν στις χώρες μέλη. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το κλειδί για την τελική εφαρμογή. Μεταξύ των όσων είπατε Λίδια, άκουσα με ικανοποίηση ότι θέλετε να ληφθεί υπόψη η κατάσταση των Ρωμά και στις ε, υποψήφιες χώρες. Πολύ σημαντικό αυτό. Και να δούμε αν ίσως αυτό χρειάζεται κάποιες τροποποίησεις στο κείμενο, δηλαδή να ε, εξαρθεί περισσότερο. Διάβασα με προσοχή. Άκουσα τη συνάδελφο Γιαρόκα και την ε, ευχαριστώ και για την ε, διάβια και για τη σαφήνεια με την οποία εκφράστηκε. Έχω μερικές σκέψεις όμως να πω. Εντάξει για τη στρατηγική ένταξης, εντάξει για τις ε, προτεραιότητες. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μία χαρτογράφηση των κρατών μελών. Χρηματοδοτήσεις. Στα τέλη Σεπτεμβρίου η κυρία Ρέντινγκ μας είπε ότι δημιούργησε μία task force που σύντομα μέχρι τον Απρίλιο θα μας είχε δώσει συγκεκριμένα ε, αποτελέσματα για τη χρήση των κονδυλίων ε, εκ μέρους των κρατών μελών. Διότι όπως είπε και η κυρία Γιαρόκα, η χρήση αυτών των κονδυλίων αποτελεί ένα σημαντικό τμήμα του όλου σχεδίου παρέμβασης. Λοιπόν, αυτό το σχέδιο είναι ένα σχέδιο συμπερίληψης. Μπορεί να μας δώσει τη δυνατότητα, αν πετύχει, να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου είδου σχέδια και σε άλλες πραγματικότητες. Οπότε ένα τέτοιο σχέδιο μπορεί να εφαρμοστεί μετά συνολικά και σε ένα άλλο σχέδιο για τους μετανάστες για παράδειγμα διότι όπως είπε και η συνάδελφος, όπως είπε και η συγγήτρια, είναι πολύ σημαντική η αλληλεγγύη. Θα πρέπει πριν ολοκληρώνω να γίνει η αναφορά στους νέους και στην κατάρτιση των νέων όπως επίσης και το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής της κατάρτισης για τους νέους. Ο κύριος Μπέλντερ. Ευχαριστώ. Και εγώ βρίσκω πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία στην έκθεση και θα την υποστηρίξω. Σε πολλές ακροάσεις έχω ακούσει το θέμα της χρηματοδότησης, δηλαδή πόσα κονδύλια έχουν δοθεί. Γίνεται λόγος για 1,4-1,6 δις σε σχέση με τα συνολικά κονδύλια όταν ρώτησα πώς έχουν δαπανηθεί αυτά τα χρήματα. Δώστε μου ένα καλό παράδειγμα δαπάνης και έγινε λόγος για ένα ε, project στην Ουγγαρία ένα project διαλόγου στην Ουγγαρία, έτσι μου ελέγχθη. Θα ήθελα όμως γενικότερα να ξέρω ποιες είναι οι επιτυχίες, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε συστάσεις για το μέλλον. Και θα ήθελα να διερευνήσουμε λίγο περισσότερο αυτή την πτυχή του θέματος, για να δούμε πώς μπορούμε να κινηθούμε επιτυχώς. Ε, Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Γιαρόκα για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι έχει μεγάλη σημασία να επαναλαμβάνουμε διαρκώς ότι θα πρέπει να ε, υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα αφορά πάνω από 12 εκατομμύρια ανθρώπους έκθεση δεν είναι ιδιαίτερα πολιτική, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την γαλλική πολιτική που απομάκρυνε πολλούς πολίτες από τη χώρα και αυτή την πολιτική να την βάλουμε επί χάρτου. Νομίζω ότι τα περισσότερα σημεία είναι σωστά. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Ε, ένα γενική υφίστεμα αφορά την ε, ενσωμάτωση των Ρωμά και ήταν ένα θέμα της ακρόασης. Μιλήσαμε και για την κοινωνική ένταξη. Συμφωνώ και με τον κύριο Μολούντερ σε σχέση με την αξιολόγηση. Θα πρέπει να προβούμε σε μία αξιολόγηση του τι έγινε μέχρι τώρα, διότι έχουν χρησιμοποιηθεί πολλά χρήματα, αλλά τα χρήματα δεν ε, χρησιμοποιήθηκαν εκεί που θα έπρεπε. Και εάν δεν εντοπίσουμε τα πράγματα σωστά, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη για το μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η Ρωμά είναι μία ομάδα ανθρώπων που δεν εκπροσωπείται επαρκώς στα διάφορα κυβερνητικά σχήματα ή όργανα και αυτό θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς. Άρα οι Ρωμά μπορούν να είναι ο αποδιοπομπαίος τράγος των πολιτικών των κρατών μελών. Θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στη λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον. Η κυρία Γκυγιόμ. Να συγχαρώ και εγώ την κυρία Γερόκα για τη δουλειά της που είναι πάρα πολύ θετική. Πρόκειται για μία ισορροπία η οποία δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο να προσεγγιστεί και να υλοποιηθεί διότι φύγει και άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν με θέματα παινίας κλπ. Στο προηγούμενο κείμενο είχαμε συζητήσει και επιμείνει για μια στρατηγική που να διαρθρώνεται σε όλα τα επίπεδα. και στις χώρες προέλευσης και στις χώρες υποδοχής. Νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερες προτάσεις που συνδέονται με τη χώρα προέλευσης και όχι με εκείνη υποδοχής. Συμφωνώ λοιπόν με τη συνάδελφο Μποσκούτ να ληφθούν ε, ε, ε, κάποια μέτρα και για τις χώρες υποδοχής των Ρώμα. Φαντάζομαι ότι με τις τροπολογίες μας θα παρέμβουμε για να τα αλλάξουμε τα πράγματα. Τώρα προσέξτε, επειδή εγώ επιμένω πολλές φορές με την ορολογία. Ε, στα γαλλικά γίνεται αναφορά για παθητικότητα, εχθρότητα και ρατσισμό κατά των τσιγκάνων. Παρακαλώ να προσέξετε όλους αυτούς τους όρους, οι οποίοι αποδίδονται δύσκολα στις διάφορες γλώσσες. Κυρία Βίκτρομ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την εργασία την οποία επιτελεί. Πιστεύω ότι το θέμα των Ρωμά αφορά πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Τώρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε πραγματικά ουσιαστικά προγράμματα δράσης σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και ένα σχέδιο Μάρσαλ για τους Ρωμά. Σε όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουμε μία ολιστική προσέγγιση όταν μιλάμε για κοινωνική ένταξη η, η έτσι ακριβώς το αντιμετώπισε το ζήτημα παραθέτοντας όλες τις πτυχές του θέματος. Υπάρχουν όμως στοιχεία που λείπουν. Δεν γίνεται καμία μνήα στα ψηφίσματά μας υπέρ των Ρωμά, ούτε στο, στις εκδιώξεις από την Γαλλία και την Ιταλία. Αυτό το θέμα θα πρέπει να αφηγεί, σύμφωνα με την έκθεση ένα άλλο βασικό βήμα είναι να ξέρουμε τι έγινε στο παρελθόν. Αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας, δεν υπάρχει μέλλον και θα περιοριστούμε στην παρούσα κατάσταση. Θα πρέπει να δούμε ιστορικά πώς εξελίχθηκε η κατάσταση των Ρωμά σε όλα τα κράτη-μέλη. Ένα σημείο εκκίνησης θα ήταν να διαδώσουμε αυτή την έκθεση μέσω και, της, ε, και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά σε αυτή την ε, απάνθρωπη κατάσταση. Για να φτάσουμε στους στόχους μας θα πρέπει να, ε, να στραφούμε προς την ιστορία. Επίσης θα πρέπει να τονίσουμε στα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση για όλους τους ε, πολίτες της Ευρώπης και δεν γίνεται καμία μνήα σε αυτή την έκθεση στην ε, ελεύθερη διακίνηση των πολιτών. Η ελεύθερη διακίνηση είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κανένας δεν θα πρέπει να αποκλείεται από αυτή την πολιτική. Πρόκειται για ένα πολιτισμικό ζήτημα. Πώς ε, μεταχειριζόμαστε τους ανθρώπους στις κοινωνίες μας τον 21ο αιώνα. Και αυτό είναι και το βασικό μου μήνυμα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την διεξοδική αυτή εργασία και σας παρακαλώ να λάβετε υπόψη τα, τα ευρωπαϊκά ψηφίσματα, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου όταν προωθείτε αυτή την εργασία. Σας ευχαριστώ για όλες ε, τις ε, συνεισφορές και για αυτές που δεν έφτασαν στο σχέδιο. Η κυρία Γερόκα θέλει να απαντήσει, η οποία μιλάει. Θέλετε να σχολιάσετε τα όλα όσα ακούσαμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να λάβω το λόγο εντάχει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα σημαντικά θέματα και θα λάβω υπόψη και τις πρωτολογίες διότι είμαστε περιορισμένοι ως προς το κείμενο. Τόσο μεγάλο θα μπορούσε να είναι το κείμενο, γι' αυτό ε, έχω εισαγάγει και έχω εντάξει όλα τα σημεία που μπορούσα. Δηλαδή είμαστε κάπως περιορισμένοι, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ενταχθούν όλα τα θέματα που θίξατε. Κυρία Βέμπερ, σκιώδης, η σκιώδης εισηγήτρια, μίλησε για το θέμα του χρονισμού και το κατά πόσο θα μιλήσουμε για μια εθνική πλαισίωση. Συντάσσω αυτή την έκθεση για ακριβώς αυτό το λόγο, διότι η Ουγγρική Προεδρία ήταν η μόνη η οποία είχε ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα και αναμένει τη χνομοδότηση του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή επίσης βασίζεται σε αυτή την έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γι' αυτό νομίζω ότι πριν από τον Απρίλιο θα πρέπει να είναι έτοιμη αυτή η έκθεση έτσι ώστε να την χρησιμοποιήσει η Κομισιόν. Άρα σε αυτό το έγγραφο ζητούμε ένα πρόγραμμα δράσης μέχρι τον Απρίλιο έτσι ώστε μέσα σε τρεις μήνες να το συζητήσει το θέμα το Συμβούλιο και τον Ιούνιο να εκκινήσει αυτή η πολιτική μέσα στα πλαίσια μιας πραγματικής δράσης που έχουμε ζητήσει και ζητούμε εδώ και έξι χρόνια. Δέχομαι αυτά που είπε η κυρία Έρνστ σε σχέση με τους ανηλίκους και τις χώρες ε, διεύρυνσης. Θα πρέπει να ενταχθούν μέσω τροπολογιών και θα το κάνω εγώ αυτό αν δεν το αναλάβει κανένας άλλος. Νομίζω ότι θα συντάξουμε πολύ καλά το κείμενο. Ε, αν δεσμεύονται τα κράτη-μέλη, πώς δεσμεύονται ως, την, ως προς την ελεύθερη διακίνηση, δηλαδή το ψήφισμα υπέρ των Ρωμά που ε, εγκρίναμε πρόσφατα. Υπάρχουν πολλά έχοντας υπόψη για να δείξω ότι υπάρχει ε, ένα νήμα που διέπει όλο μας, ολόκληρο το σκεπτικό μας και τα θεσμικά όργανα λένε το ίδιο ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή στρατηγική υπέρ των Ρωμά. Υπ' αυτή την έννοια οι εκπρόσωποι των πολιτών έχουν ψηφίσει υπέρ του ζητήματος αυτού, θα πρέπει να φτάσουμε σε μια δεσμευτική, στη δεσμευτική εξέλιξη αυτής της ε, πρότασης, όπου δεν θα μπορέσουν να υπεκφύγουν τα κράτη-μέλη, γιατί πρόκειται για ευθύνη των κρατών μελών. Και τι μπορεί να είναι επιτυχές σε τοπικό επίπεδο. Άρα δεν θέλουμε να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά τα κράτη-μέλη. Υπάρχει αυτή η στρατηγική έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να ανταποκριθούν ως προς τις δεσμεύσεις τους. Άρα αυτά που είπε ο η κυρία Μίλντερ και η Γιακολίνο είναι πολύ σημαντικό, καθώς και η κυρία Μπόσκορτ για το πώς θα δαπανηθούν τα χρήματα. Η Κομισιόν έχει προβεί στη σύσταση μιας task force Άρα ήδη μέχρι το Δεκέμβριο θα δούμε πώς έχουν λαπανηθεί τα κονδύλια από τα κράτη-μέλη. Ορισμένοι λένε ότι κανείς δεν έχει, ότι μερικές χώρες δεν έχουν ζητήσει χρήματα για την κοινωνική ένταξη. Και θα δούμε πού και πώς δαπανήθηκαν τα χρήματα ή αν έγινε κακοδιαχείριση. Άρα η έκθεση της Επιτροπής το Δεκέμβριο θα είναι ακρογωνιαίος λίθος της πολιτικής μας. Επίσης τον Απρίλιο θα έχουμε μία πρόταση για μία στρατηγική υπέρ των Ρωμά. Άρα για την Task Force θα ήθελα να την κρατήσουμε ως συντονιστικό όργανο αυτής της στρατηγικής. Επίσης μιλάμε για την πρόορη εγκατάλειψη του σχολείου από αυτά τα παιδιά. Η κυρία Ρέντιν θα συντάξει μια έκθεση που θα ανακοινωθεί το Φεβρουάριο για να δούμε κατά πόσο μπορούμε να σταματήσουμε με την ξεχωριστή εκπαίδευση στην Ευρώπη. Η κυρία Μπόσκορτ και η κυρία Βίσερ είπαν κατά πώς θα πρέπει να έχει πολιτικό χαρακτήρα αυτή η έκθεση και ποια είναι η ανθρώπινη διάσταση της έκθεσης. Είδαμε πολλά ψηφίσματα αλλά και πληθώρα ε, παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλές ε, στιγμές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η οδηγία θα μπορούσε να επιλύσει πολλά θέματα. Άρα, μέχρι το πρόγραμμα δράσης τον Απρίλιο, θα ήταν σκόπιμο να δούμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παραβίαση, συμμόρφωση, ε, δαπάνη κονδυλίων. Θα πρέπει να μάθουμε κατά πόσο οι Ρωμά γνωρίζουν τι διακρίσεις υφίστανται Άρα θα δούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτης γενεάς και μετά δεύτερης και τρίτης. Θα πρέπει να πιέσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να έχουμε οργανώσεις Ρωμά να ε, χρηματοδοτούνται και να μην χειραγωγούνται πολιτικά. Δηλαδή να αποκτήσουν μεγάλη, μεγαλύτερη δύναμη οι Ρωμά και το θέμα της ηγεσία θα πρέπει να μας απασχολήσει. Μας ενδιαφέρει και το ιστορικό της υπόθεσης. Γιατί η παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων προέρχεται από το γεγονός ότι δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας είχαμε κοινή εκπαίδευση, αλλά ε, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε υπό τα κομμουνιστικά καθεστώτα. Δηλαδή, μαθαίνουμε η μεν για τους δε μέσω των ΜΜΕ ή από τραγωδίες. Έχει μεγάλη σημασία τα σχολικά προγράμματα να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική ζωή, κοινωνική ζωή των μειονοτήτων και για τον Ιανουάριο, για την Ολομέλεια, να λάβουμε υπόψη ε, ένα κοινό σχέδιο αντιμετώπιση των Ρωμά, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσοι Ρωμά σκοτώθηκαν ε, ή ε, χάθηκαν στα, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη όλες τις μειονότητες που έχουν συνεισφέρει οικονομικά και κοινωνικά και που σήμερα συνεισφέρουν. Γιατί οι Ρωμά συνεισφέρουν και οικονομικά. Ακόμα και στην παράνομη εργασία, διότι υπό κομμουνιστικά καθεστώτα το 98% των Ρωμά ε, ασχολούνταν, δηλαδή απασχολούνται με επίσημη εργασία. Ενώ τώρα υπάρχει ένα 12% μόνο των Ρωμά που απασχολούνται επίσημα. Όλοι οι άλλοι είναι παράνομοι. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την εισηγήτριά μας και εδώ νομίζω συνοψίζεται πια η συζήτηση, ολοκλώνεται η συζήτηση σε αυτή την φάση του σχεδίου εκθέσεως. Υπενθυμίζω την προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 10 Ιανουαρίου, Δευτέρα, στις 12. Και η επόμενη φάση θα είναι τις 3 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Ευχαριστούμε κυρία Γιαρόκα λοιπόν και πάλι και αναμένουμε με ενδιαφέρον την περαιτέρω πορεία του θέματος αυτού που συνδέει την Επιτροπή ε, Θεμελιδών Ευθεριών με την Επιτροπή Απασχολήσεως. Προχωρούμε στο επόμενο θέμα της ε, ημερησίας <coughs> διατάξεως. Γνωρίζετε ότι τα 7 και 8 έχουν αναβληθεί. Προχωρούμε λοιπόν στο 9. που φέρει τον τίτλο «Δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Εδώ παρούσα είναι η κυρία Μπίργκιτ Ζίπελ, η συγγήτρια. Εν πάση περιπτώσει σε αυτή την φάση της συζητήσεως αυτά που έχουμε είναι από ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τα δικαιώματα υπόπτων σε ποινικέ διαδικασίες να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και για τις ε, κατηγορίες που τους ε, απαγγέλλονται. Έχει γίνει η προσαρμογή από το Συμβούλιο το Νοέμβριο του 2009 και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το πρώτο βήμα περατώθηκε επιτυχώς τον Ιούνιο του 2010 με συμφωνία επί της οδηγίας για δικαιώματα μεταφράσεως και διερμηνία σε ποινικέ διαδικασίες. Το Συμβούλιο κατέληξε σε κοινή θέση επί της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 3 Δεκεμβρίου. Τώρα έχει, έχει έρθει η σειρά του Ευρωκοινοβουλίου να ε, καταλήξει σε θέση για να προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με το Συμβούλιο. Θα ακούσουμε τώρα την εισηγήτριά μας κυρία Μπίρκιτ Ζίπελ και μετά θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση. Νομίζω ότι η Επιτροπή είναι παρούσα και επίσης μπορεί να ακουστεί και η φωνή του Συμβουλίου. Πρώτα όμως η κυρία Ζίπελ. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σε αυτή την πρώτη παρουσίαση του θέματος να περιοριστώ στα πλέον σημαντικά στοιχεία. Μιλούμε για μια νέα Ευρώπη και με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης μιλούμε και για τη δημιουργία ενιαίου χώρου δικαίου. Ωστόσο μέχρι τώρα έχουμε 27 πολύ διαφορετικά νομικά συστήματα και εδώ οι πολίτες αξιώνουν ταχείες αλλαγές. Στο παρελθόν είχαμε ρίξει ιδιαίτερο βάρος στην συνεργασία μεταξύ των αρχών για το θέμα αυτό. Σε τότε τότε την ε, οδηγία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μπαίνει ο πολίτης και τα δικαιώματά του εφόσον εμπλέκεται σε ποινική διαδικασία. Και νομίζω ότι ορθό θα είναι να διασφαλίσουμε δίκαιη διαδικασία σε ολόκληρη την Ευρώπη σύμφωνα και με, τις, ε, με την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Εν προκειμένου σημαντικά είναι τα διαδικαστικά δικαιώματα η διαβούλευση με συνήγορο, η, το δικαίωμα μετάφρασης και διερμηνίας. Αυτό που έχουμε τώρα μπροστά μας είναι το δικαίωμα της ενημέρωσης, της πληροφόρησης, διότι μόνον όποιος γνωρίζει ποια δικαιώματα διαθέτει μέσα σε μια ποινική διαδικασία μπορεί πράγματι να τα αξιώσει, να αξιώσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών. Επίσης δε, η μη λήψη υπόψη από πλευρά των αρχών των δικαιωμάτων αυτών σημαίνει θέση σε κίνδυνο του δικαίου της διαδικασίας. Για το λόγο αυτό χαίρομαι για την υποβληθήσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θεωρώ ότι πρόκειται για μια πραγματικά ε, ορθή βάση για την περαιτέρω συζήτηση. Οι τροποποίησεις που σκέπτομαι να ζητήσω για την πρόταση της Κομισιόν κινούνται κυρίως προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ώστε η οδηγία να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στέρησης των ελευθεριών, ακόμη και αν δεν εφαρμόζονται όλα τα δικαιώματα σε όλες τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, αν συλληφθώ εγώ ως Γερμανίδα στη Γερμανία, δεν έχω ανάγκη από διερμηνία και μετάφραση. Αλλά θα πρέπει όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στη δική μου περίπτωση, στη δική μου ε, κατάσταση, να έχουν όλα αυτά τα δικαιώματα. Θα προτείνω επίσης τα ελάχιστα δικαιώματα του άρθρου 3 να διευρυνθούν τουλάχιστον με συμπερίληψη του δικαιώματος σιγής, σιωπής. Και θέλουμε επίσης και σε περίπτωση συλλήψεως να περιλαμβάνονται στην ενημέρωση και άλλα δικαιώματα όπως για παράδειγμα η διάρκεια της ε, κράτησης για την προανάκριση. Αυτά πρέπει όχι μόνο να μπορεί να τα διαβάσει ο ενδιαφερόμενος, αλλά και να τα κρατήσει. Και όσοι για παράδειγμα δεν μπορούν να διαβάσουν καλά διότι ίσως έχουν προβλήματα όρασης, αλλά επίσης και ανήλικοι οι οποίοι έχουν ανάγκη από εξηγήσει. Είναι αυτονόητο το ερώτημα ότι ο κατηγορούμενος θα πρέπει να ενημερώνεται ακριβώς για Ποιε κατηγορίες το απευθύνονται, το απαγγέλλονται. Είναι απαραίτητο επίσης να έχει και πλήρη πρόσβαση σε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχέ και αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Τελειώνοντας θα επισημάνω το εξής. Θα προτείνω δηλαδή στην Επιτροπή η επιστολή υπόδειγμα που βρίσκεται στο παράρτημα θα πρέπει να είναι δεσμευτική, υποχρεωτική, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφέ. Βεβαίως, κάθε χώρα μέλο θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να προσφέρει παραπάνω δικαιώματα στον ε, κατηγορούμενο. Κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνοντας, εκφράζω τη λύπη μου ρητά για το ότι δεν κατέστη δυνατόν να ψηφιστούν όλα τα διαδικαστικά δικαιώματα σε μία ενιαία διαδικασία. Και είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν τώρα να προχωρούμε βήμα-βήμα, να συζητούμε δηλαδή ένα διαδικαστικό δικαίωμα μετά το άλλο και αυτό είναι λυπηρό διότι με τον τρόπο αυτό η βελτίωση των ελάχιστων προδιαγραφών των διαδικαστικών δικαιωμάτων υπέρ των πολιτών θα αρχίσει να γίνεται ορατή στα μάτια των πολιτών μόνο μετά από πάροδο πολλών ετών. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν με την ευκαιρία Θα ευχαριστήσω την συνεργάτη μου η οποία έχει εργαστεί πολύ. Θα ευχαριστήσω και την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και βεβαίως με μεγάλη μου χαρά θα ακούσω ήδη σήμερα όσο το δυνατόν περισσότερα σχόλια και προτάσεις των συναδέλφων μου για να μπορέσω να εκπονήσω περαιτέρω το κείμενό μου. Ο πρόεδρος, ωραία. Ας ακούσουμε τώρα τον εκπρόσωπο ή την εκπρόσωπο της Επιτροπής και μετά τη Βελική Προεδρία του Συμβουλίου. Κύριε Α, η κυρία πρώτα από τη Βελγική Προεδρία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω να μιλήσω εδώ εξ ονόματος της Βελγικής Προεδρίας. Το σχέδιο οδηγίες υποβλήθηκε στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 3 Δεκεμβρίου και έγινε μία αρχική εξέταση από το Συμβούλιο εκτός από τα παραρτήματα, δηλαδή διατάξεις και εκτιμώντας. Η συμφωνία που, στην οποία καταλήξαν εδώ και μερικού, σε λίγους μήνες αποδεικνύει το ενδιαφέρον που τρέφουν τα κράτη-μέλη για το δικαίωμα της υπεράσπισης. Απ' την άλλη μεριά υπήρχε μια δυσκολία του να αντικατοπτριστούν μέσα στη διάταξη όλες οι ένομες τάξεις των κρατών μελών. Οπότε διαμορφώσαμε μια συνένεση. Παραμένει όμως η βασική ανησυχία της ε, διαφοράς ε, των ενόμων τάξεων των κρατών ε, μελών ε, και των συστημάτων. Τώρα η σκητάλη θα περάσει στην Ουγγρική Προεδρία που ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσει τις συζητήσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για αυτήν τη γρήγορη συμφωνία είναι ουσιαστικό να κρατήσουμε την δυναμική για αυτό το ντοσιέ των διαδικαστικών εγγύσεων εγκρίνοντας το πρώτο μέτρο της roadmap που ήταν ουσιαστική για να διατηρήσουμε τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων μέτρων της roadmap και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις ε, διαδικαστικές εγγύησεις και τα δικαιώματα των ανθρώπων σε αυτό τον τομέα. Ευχαριστώ. Η Κομισιόν. Ευχαριστώ, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομη. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κυρία Σίπελ για τα θερμά της λόγια λάβαμε το σχέδιο έκθεσης σήμερα και ρίξαμε μία πρώτη ματιά, δεν το έχουμε αναλύσει εις βάθος, αλλά εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμφωνήσουν, κάτι το οποίο είναι ιδιαίτερα θετικό. Επίσης με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να πω ότι είναι ευπρόσδεκτη η προσέγγιση του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου εξαιτίας των προσπαθειών της Βελικής Προεδρίας και υπό την Προεδρία της Μαρία Ελέν Χέα και ελπίζουμε να προχωρήσουμε στον τριμερή διάλογο το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Τώρα ας δώσουμε το λόγο στα μέλη. Ο κύριος um, Μπουζούτιλ. Θα ήθελα να λάβω το λόγο ε, εξ ονόματος του κυρίου Αντωνέσκου και άλλων συναδέλφων που υπέβαλαν τις απόψεις τους. Ε, δυστυχώς δεν βρίσκεται κανένας μαζί μας. Γι' αυτό θα υποβάλω τα σχόλιά τους. Θα ήθελα να ε, εκφράσω την υποστήριξη του ε, προς αυτή την οδηγία και επειδή ασχοληθήκαμε με αυτό τον τομέα που είναι ε, μεγάλη σημασία, όπως είπε και η συγγήτρια, ίσως θα ήταν καλύτερα να είχαμε διαφορετική προσέγγιση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε και θα αρκεστούμε σε αυτήν. Εντάχει τώρα να δούμε τα επιμέρους ζητήματα που το ΕΛΚ θα ήθελε να θίξει ως προς το άρθρο 3 σε σχέση με τον κατηγορούμενο ο οποίος ε, θα πρέπει να, ε, στον οποίο θα πρέπει να δοθούν οι σωστές πληροφορίες θα πρέπει να πούμε ποιες αρχές θα χορηγήσουν αυτές τις πληροφορίες και πώς θα γίνει αυτό. Γραπτός προφορικά το ίδιο αφορά και το άρθρο 6 που αναφέρεται στο δικαίωμα πληροφόρησης σε σχέση με το κατηγορητήριο. Στο άρθρο 3, θέλουμε περισσότερες ε, διατάξεις τη στιγμή που ο υπόδικος είναι ανήλικας όπως ήδη ελέγχθη ή εάν δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τις ε, πληροφορίες που του παρέχονται πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται ανάλογα με τις ανάγκες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πολιτών. Σε σχέση με το άρθρο 8, θα θέλαμε οι εκπρόσωποι της Επιτροπής, της Επιτροπής να μας πει περισσότερα πράγματα ως προς τη διαδικασία και ποια είναι η πλέον ενδεδειγμένη για την παρούσα κατάσταση, ιδιαίτερα ως προς την αποδοχή ε, λήψη πληροφοριών από τον ενδιαφερόμενο. Ως προς το δικαίωμα στη σιωπή, συμφωνούμε με άλλους ε, συναδέλφους ότι υπάρχει αυτό το δικαίωμα μη αποκάλυψη στοιχείων, δηλαδή της σιωπή. Αυτό είναι μεταξύ άλλων δικαιωμάτων που δεν ε, συμπεριλαμβάνονται και είναι κρίμα γιατί έχουμε τονίσει ότι μέσα στα πλαίσια της δίκαιης δίκης ε, υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Ίσως αυτό αφορά έλλειψη θέλησης από ορισμένα κράτη-μέλη, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να φτάσουμε σε ένα συμβασμό για να συμπεριληφθεί και αυτό το στοιχείο. Ελπίζουμε η συγγήτρια να το δει έτσι ώστε να προτείνει ένα συμβασμό. Νομίζω ότι κάλυψα όλα τα σημεία. Υπάρχει και ένα τελευταίο σε σχέση με το ποιος ε, παρέχει τις πληροφορίες και κατά πόσο έχουν, ε, έχει το προσωπικό αυτό την ε, κατάλληλη κατάρτιση ως προς τον κατηγορούμενο, την πρώτη επαφή, δηλαδή η πρώτη επαφή μεταξύ κατηγορούμενου και, κατηγορούμενου και ανακριτή ή ενός αξιωματικού της αστυνομίας, ίσως να μην είναι η καλύτερη δυνατή επαφή και δεν θα πρέπει να έχουμε ε, κακοχρησία αυτού του μέσου. Αλλά βέβαια υπάρχουν και οι εμπλεκόμενες δαπάνες θα πρέπει να μας απασχολεί σε αυτό το θέμα γιατί το κόστος μπορεί να είναι εκρηκτικό και να επιμηκύνει τη διαδικασία. Αυτά τα ζητήματα μου ζήτησαν οι συνάδελφοι να θίξω. Μερικά τα έχει ήδη εξετάσει η συγγήτρια. Το ΕΛΚ όμως θα συνεισφέρει γενικότερα στην ολοκλήρωση αυτής της έκθεσης. Ευχαριστούμε κύριε Κύριε Βίξτρομ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω εξ ονόματος της Σάρα Λάτφορντ που είναι ισχυώδης από πλευράς φιλελευθέρων. Θα ήθελα να εκφράσω τα, τις θερμές μου ευχαριστίες προς την κυρία Σίπελ γιατί συνεργάστηκε πολύ καλά με τους σκιώδεις. Η κυρία Λάντφορτ θα ήθελε να τονίσει την υποστήριξή μας όχι μόνο ως προς τα διασυνοριακά μέτρα δίωξης, αλλά και την πρόθεση των δικαιωμάτων των ε, κατηγορουμένων, έτσι ώστε να προωθούνται δίκες ε, δίκες. Δεχόμαστε τη δεύτερη πρόταση στον οδικό χάρτη και στην οδηγία περί διερμηνίας και μετάφρασης, όπως είπε και η κυρία Λάντφορ ως εισηγήτρια, θεωρεί ότι αυτά τα δικαιώματα δεν ισχύουν όταν έχουμε να κάνουμε με ένα πλημέλημα και εάν ισχύουν οι ρήτρες διασφάλισης επίσης. Το ίδιο ανέφερε και το Συμβούλιο. Όμως δεν υπάρχει παραλληλισμός, όπως είπε το Συμβούλιο της Ευρώπης, διότι σε ορισμένες περιστάσεις ε, οι ύποπτοι για ε, μικρά, για περιορισμένα πλημελήματα θα πρέπει να έχουν δικαίωμα πληροφόρησης. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχει αποκλεισμός. Στο άρθρο 3 ως προς τον κατάλογο δικαιωμάτων και πληροφοριών το Συμβούλιο προσέθεσε και το δικαίωμα της ε, και το θέμα προσαγωγή σε δικαστήριο. Εγκαίρος θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι έγκυρες, έγκυροι αυτοί οι περιορισμοί. Συμφωνώ με την κυρία Σίπελ ως προς την ε, διευκρίνηση για τις πληροφορίες που μπορεί να λάβει ένας υπόδικος κρατούμενος, αλλά δεν θεωρώ ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να αφορούν μόνο ε, τις ε, κατηγορίες, γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά. Θα ήθελα να επιταχύνω τη διαδικασία έτσι όλοι να απολαύσουμε ένα ωραίο βράδυ. Θα ήθελα ε, δυνάμει του άρθρου 8.3 που αναφέρει ότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν γίνονται αποδεκτά στη διαδικασία αν δεν είναι παρκώς τεκμηριωμένα. Μπορεί να μας πει γιατί ισχύει κάτι τέτοιο και τι θα σήμαινε έμπρακτα τη στιγμή που θα πρέπει να δούμε το παραδεκτό των αποδεικτικών στοιχείων ε, μέχρι ότου υπάρξει μια εναρμόνιση. Επίσης δεν γίνεται μνήα στο κείμενο ως προς το δικαίωμα πληροφόρησης σε θέματα τα οποία δεν έχουν συζητηθεί από τον οδικό χάρτη. Και εδώ μιλώ και προσωπικά. Το, τα δικαιώματα αυτά αφορούν το δικαίωμα περίθαψης, εγγύησης και επαφής με κάποιο συγγενικό πρόσωπο. Ίσως θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και άλλα δικαιώματα στο μέλλον. Αυτά ήθελα να πω εξ ονόματος της Σάρα Λάντφορντ και μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Πίκστρομ. Εξαιρετική η εργασία σας. Ε, αναφέρατε αυτά που σας απασχολούν και νιώθουμε και την παρουσία της κυρίας Λάντφορντ μέσα από αυτή την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Ζίπελ για την κατά τη γνώμη μου πολύ επιτυχημένη παρουσίαση του θέματος ε, στο σχέδιό της. Δεν μιλώ εξ ονόματος μόνο των Πρασίνων αλλά και ως ε, συντάκτης γνωμοδότησης της Επιτροπής Νεότητας που ακόμα δεν έχει γνωμοδοτήσει αλλά που επιθυμεί να το πράξει πριν από την ψηφοφορία που θα διεξαχθεί εδώ στην Λίμπε τον Ιανουάριο και σας ευχαριστούμε που ε, μας λάβατε υπόψη. Για τα όσα λέχθηκαν μέχρι τώρα έχω μόνο μερικά συγκεκριμένα ε, σχόλια και ορισμένα γενικότερα. Διότι εδώ νομίζω συμφωνούμε για πολλά θέματα τα οποία εμφανίζονται και στην ανακοίνωση της Επιτροπής αλλά ίσως χρήζουν συμπληρώσεων. Για παράδειγμα, η συζήτηση για το ε, δικαίωμα να τηρήσει κανείς σιγή. Το ζήτημα επίσης να ζητήσει κανείς προξενική ε, βοήθεια. Αυτό βέβαια δείχνει ότι βρισκόμαστε μέσα σε μια διαδικασία όπου δεν πρόκειται μόνο θέμα δικαιώματος πληροφόρησης και αυτό χρειάζεται βελτίωση βέβαια αλλά και που εντάσσεται σε ένα οδικό χάρτη που πάει να εναρμονίσει τα διαδικαστικά δικαιώματα σιγά σιγά. Και αυτό είναι απαραίτητο, απόλυτα αναγκαίο. Τα τελευταία χρόνια έχουμε λάβει διάφορα μέτρα όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Συλλήψεως. το σύστημα αποδεικτικών στοιχείων. Τώρα, τα διαδικαστικά δικαιώματα των συλληφθέντων που δεν έχουν για παράδειγμα καμία ενημέρωση, καμία πληροφορία για το ποια είναι τα δικαιώματά τους. Και είναι πολύ σημαντικό σε μια τέτοια κατάσταση, ακριβώς εκεί όπου μάλιστα ακριβώς ένα χρονικό σημείο όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση πάει να μπει στην συνθήκη α, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε και την συνθήκη της Λισαβόνας που περιλαμβάνει τον χάρτη των δικαιωμάτων ως αναπόσπαστο τμήμα της. Νομίζω λοιπόν ότι και το Συμβουλίο και οι χώρες μέλη πρέπει να αντιληφθούν ότι υπάρχει αναγκαιότητα και ότι αυτή η αναγκαιότητα συνδέεται άμεσα με το ερώτημα της ενημέρωσης για τα διαδικαστικά δικαιώματα. Οι διαδικαστικές προδιαγραφές που μέχρι τώρα έχει θεσπίσει με την ομολογία του και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και που είναι δεσμευτικά για όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι σε συγκρίσιμο επίπεδο και να ισχύουν σε συγκρίσιμο επίπεδο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και να περιληφθούν σε αυτό το δίκαιο, τη ρύθμιση δηλαδή περί πληροφόρησης. Για παράδειγμα, η πρόσβαση στα διαδικαστικά έγγραφα είναι ουσιώδης. Σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες θα πρέπει να, έχουν και, να μπορούν να έχουν δηλαδή και την εμπιστοσύνη στο γεγονός δηλαδή ότι ισχύουν σε όλες τις χώρες μέλη ορισμένα ελάχιστα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουν. Αυτό που θα ήθελα εγώ θα ήταν στη συζήτηση αυτή να μην περιοριστούμε μόνο να πούμε να βρούμε κάπως στα γρήγορα και μια αιτιολόγηση για μια καλύτερη αμοιβαία αναγνώριση, αλλά πραγματικά να ξεκινήσουμε από τα κάτω και να εναρμονίσουμε τα διαδικαστικά δικαιώματα, τα οποία μάλιστα θα μπορούν να βελτιώνονται σταδιακά. Και σε αυτή την ε, Letter of Rights, σε αυτή την επιστολή δικαιωμάτων, να μπορούν να επανεξεταστούν μέσα στα πλαίσια αυτού του οδικού χάρτη που ανέφερα προηγουμένως. Να υπάρξει ίσως και μια ρήτρα ευελιξίας ότι δηλαδή εάν συμφωνήσουμε σε μια παραπέρα εναρμόνιση διαδικαστικών δικαιωμάτων να περιλαμβάνονται και αυτά σε αυτή την ενημέρωση, την υποχρεωτική ενημέρωση που θα κάνει η αρχές για τα διαδικαστικά δικαιώματα. Κατά τα άλλα δεν έχω πολλά να συμπληρώσω στην έκθεση της κυρίας Ζίπελ. Θα εγκύψει σε αυτήν η Επιτροπή μας και θα κάνουμε και εμείς μια γνωμοδότηση ίσως με κάπως διαφορετικές αποχρώσεις, αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι το Κοινοβούλιο να συζητήσει το θέμα αυτό και νομίζω ότι δεν πρέπει να δεχθούμε να ε, πιεστούμε χρονικά. Πρόκειται για θέμα λίγων εβδομάδων. Αυτό που χρειάζεται είναι μια συνεπή στάση που να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών. Και νομίζω ότι αυτό μπορούμε πραγματικά να το επιτύχουμε και με χαρά θα συνεργαστώ με την εισηγήτρια αλλά και με τους άλλους ε, σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ κύριε Άλμπρεχτ. Ο κύριος Τενταφυλίδης. Ευχαριστώ. Λίγα λόγια για να πω ότι και εμείς ε, συμφωνούμε με την πρόταση και με την ταχύτητα τα σύνταξης της έκθεσης από την κυρία Σίπελ. Θα ήθελα να την ευχαριστήσω. Νομίζω ότι θα πρέπει να ε, έχουμε, να έχουμε ελάχιστες νομικές προδιαγραφές σε όλες τις χώρες και συμφωνώ με αυτά που είπε η κυρία Σίπελ ότι η πρότυπη επιστολή θα μπορούσε να εγκριθεί από τα κράτη-μέλη. Συμφωνούμε με τις περισσότερες τροπολογίες που έχει ήδη υποβάλει και θα υποβάλουμε και τις δικές μας Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία που ίσως θα μπορούσαν να βελτιωθούν, δηλαδή η υπόδειξη να ε, προσαχθεί κανείς άμεσα στο δικαστήριο, δηλαδή αμελητή. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σίπελ. Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή την οδηγία τάχιστα όπως κάναμε και με την οδηγία για δικαίωμα μετάφραση, μετάφραση και διερμηνία για να προχωρήσουμε με τον οδικό χάρτη Βίλαντ. Ευχαριστώ. Πριν από λίγες εβδομάδες είχα αλλάξει επιτροπή Είμαι όμως σκιώδης συγκεκριτής στην Νομική Επιτροπή και με την ευκαιρία που βρίσκομαι εδώ θα ήθελα να πω λίγα λόγια. Χαίρομαι πρώτα που η συγγήτρια κινήθηκε με τέτοια ταχύτητα. Βέβαια, εάν δεν υπάρχουν οι μεταφράσεις, εάν τρεις ημέρες πριν δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να συζητηθεί, στην ουσία μπαίνουμε εμείς οι ίδιοι σε πίεση χρόνου και το θέμα είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Δεύτερο, αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε σαφώ είναι τι ακριβώς θέλουμε. Η έκθεση αυτή είναι σχετικά απλή, εάν, ή θα ήταν σχετικά απλή, αν θέλαμε απλώς να διασφαλίσουμε ότι με την ενημέρωση αυτή περιγράφεται το τι ισχύει σε κάθε χώρα μέλος. Ότι ο, ο διότι έτσι πρέπει να χαρακτηριστεί, θα γνωρίζει ποια δικαιώματα έχει σε ποιε χώρε θα αρκούσε. Διότι αν έχουμε ένα, για παράδειγμα, Γερμανό ύποπτο, ο οποίο ανακρίνεται στη Μεγάλη Βρετανία, μπορώ να του πω, άκου το φίλε, στη χώρα αυτή, εάν σιωπήσεις, ερμηνεύεται αρνητικά. Ενώ εάν ένας Βρετανός πάει στη Γερμανία και συλληφθεί εκεί, μπορώ να τον ενημερώσω, κοίταξε να δεις, εδώ στη Γερμανία μπορεί και να σιωπήσεις, χωρί αυτό να ερμηνευθεί αρνητικά. Αυτό θα αρκούσε και θα μπορούσαμε μετά να πούμε α, πώς θα τα εναρμονίσουμε από εδώ και μπρος. Αλλά νομίζω η συζήτηση στρέφεται εδώ γύρω από το πώς θα ενημερώσω και εδώ είναι σωστό να συζητήσουμε πραγματικά και για διαδικαστικά δικαιώματα. Εάν αυτός είναι ο στόχος μας, τότε έχουμε κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα. δεν αρκεί μονάχα να ακούσει τα πράγματα αυτά. Ο υποπτό πρέπει και να τα κατανοήσει. Ούτε σημαίνει ότι ο καθένας έχει σπουδάσει νομικά ή πρέπει να έχει σπουδάσει νομικά για να μπορέσει να καταλάβει τα πράγματα αυτά. Και αυτοί που είναι, εν πάση περιπτώσει, και λιγότερο ευφύς, κάποια στοιχεία γνωρίζουν από την κοινωνικοποίηση του συστήματός του δικαιικού συστήματος μέσα στην χώρα τους. Οι άλλοι που προέρχονται από άλλες χώρες πρέπει να γνωρίζουν το αν είναι κανείς αθώος ή ένοχος είναι διαφορετική υπόθεση. Για τους ανθρώπους λοιπόν αυτούς αυτό που θα βοηθήσει εν τέλει, που θα συμβάλλει εν τέλει είναι μοναχά η εναρμόνιση. Οι χώρες μέλη λοιπόν πρέπει να αποφασίσουν επιτέλους αν θα αρκεστούν στα λόγια με διάφορες ρήτρες opt-out ή opt-in ή αν είναι διατεθειμένες να κινηθούν περαιτέρω. Βρίσκω ότι σε ορισμένους τομείς υπάρχει δυνατότητα να αναζητηθούν κάποιοι συμβιβασμοί. Σε άλλους τομείς βλέπω να είναι πολύ περιορισμένο το ενδεχόμενο αυτό. Δηλαδή βλέπω λίγες δυνατότητες συμβασμού στο πώς ερμηνεύεται η σιγή ενός αθώου ή ενός ενόχου. Επίσης πρέπει να απολυθεί από τα κρατητήρια πριν να τον δικαστής. Πάλι εδώ οι διαφορετικές νομικές παραδόσεις είναι διαφορετικές. Λέμε ότι γενικά η αστυνομία πρέπει να έχει στη διάθεσή της μια εργάσιμη ημέρα πριν να προσαχθεί στον δικαστή. 24 ώρες δηλαδή. Μπορούμε ίσως να συμβαστούμε και να πούμε 24, 36, 48 ώρες. Είναι μικρές εδώ σχετικά οι διαφορές. Επίσης πρέπει να θέσουμε και θέματα οριοθετήσεων που σε ορισμένες χώρες είναι πολύ σημαντικές. Τι γίνεται όταν κάποιος έχει ακουστεί ως μάρτυρας και μετά από την δέκατη εξέτασή του ως μάρτυρα αρχίζει και έχει κάποιες υποψίες η αστυνομία. Πού βρίσκεται λοιπόν το όριο, η κόκκινη γραμμή ας πούμε αν θέλετε. Πώς λοιπόν από ύποπτος πάει και γίνεται κατηγορούμενος. υπάρχουν και άλλες νομικές παραδόσεις που λένε σε είχαμε ως τώρα μέχρι ύποπτο θα σε αφήσουμε σε αυτήν την κατάσταση γιατί δεν υπάρχει διαδικασία που να προβλέπει κάποια συνέχεια. Εγώ πρέπει να μπορώ να κάνω την αίτηση να θεωρηθώ κατηγορούμενος και τότε θα πρέπει να κρίνει ο δικαστής εάν η κατηγορία τελικά στέκεται ή απορρίπτεται. Και αν απορριφθεί η κατηγορία τότε είμαι αθώος με πιστοποιητικό. Ας πούμε. Έχουμε λοιπόν θέματα όπως fair trial, habeas corpus, και βλέπετε και πόσο αλλάζει με την ψηφιακή τεχνολογία ο κόσμος. Ε, τα πράγματα λοιπόν, το κάθε πράγμα πόσο μένει μέσα, ε, η κάθε πράξη πόσο μένει μέσα στα ε, ψηφιακά αρχεία. Όποιος λοιπόν είναι αθώος πρέπει να έχει και το δικαίωμα να αξιώσει να αναγνωριστεί ως αθώος. Ή εάν έχει αν έχει υπάρξει υποψία σχετικά με την, με την, ε, με την αθωότητά του, θα πρέπει να μπορεί να λευκανθεί. Επίσης, πού πρέπει να ενημερώσω έναν συνήγορο ότι την επόμενη μέρα γίνεται ακροματική διαδικασία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ περίπλοκα τα πράγματα και δεν αισθάνομαι καθόλου καλά μέσα σε αυτόν τον καλπασμό που ε, προχωρούμε. Με τον κύριο Άλμπρεχτ έχω ήδη συζητήσει μία φορά και βρισκόμαστε κοντά. Εγώ είπα και στον κύριο Άλμπρεχτ να τα πει και στην ομάδα του. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον ξέφρενο καλπασμό και μείνουν left over, τα οποία τελικά θα καταλήξουν στην Ολομέλεια ως θέματα λεπτομέρειας, τότε στην πραγματικότητα υποσκάπτουμε την δουλειά που θα πρέπει να γίνει στην Ολομέλεια. Αυτά ήθελα να πω για την ώρα. Ευχαριστώ. Θα στραφούμε στην εισηγήτρια. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, δεν βλέπω άλλα σχόλια από, από μέλη, από τα μέλη μας. Η κυρία Σίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ ιδιαίτερος τον τελευταίο αγορητή που μου δίνει την ευκαιρία να επισημάνω το εξής. Πρώτο, θεωρώ και εγώ ότι όντως χρειαζόμαστε εναρμόνιση επιγόντως σε πολλούς τομείς και οι πολίτες είναι απογοητημένοι από την Ευρώπη διότι ακόμα η Ευρώπη που έχουμε είναι πολύ λίγη σε πολλούς τομείς. Προφανώς υπάρχει όμως μια παρανόηση και εγώ είπα στην αρχή πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε ταυτόχρονα όλα τα διαδικαστικά δικαιώματα αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρούμε σε διαδοχική σειρά. Και ε, συζητούμε, πάμε να εγκρίνουμε τώρα την ενημερωτική επιστολή πριν να έχουμε συζητήσει όλα τα δικαιώματα. Με αυτό λέμε μοναχά ωστόσο ότι ενημερώνουμε. Δεν εναρμονίζουμε όμως απολύτως ουδέν δίκαιο. Εάν γράψουμε στην ενημερωτική επιστολή. Και αν, το γράψω, αν γράψω λοιπόν ότι έχεις δικαίωμα ύποπτε να προσλάβει συνήγορο. Δεν σημαίνει καθόλου εναρμόνιση. Δεν υπάρχει εναρμόνιση από ποια στιγμή και μετά μπορεί να ε, έχει συνήγορο. Ποιο φροντίζει να του βρει συνήγορο. Αυτά όλα μένουν ανοιχτά. Με την παρούσα διηγεία το μόνο που εγκρίνουμε είναι η παροχή πληροφόρηση, η οποία πράγματι από χώρα σε χώρα θα είναι διαφορετική. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα, το οποίο εξήγησα στην αρχή, ότι θα ήταν πολύ καλύτερα όλες αυτές οι διαδικαστικές οδηγίες, όλα αυτά τα δικαιώματα να συζητηθούν ταυτόχρονα. Ωστόσο, δυστυχώ δεν μπόρεσε να περάσει την άποψη αυτή η Κομισιόν και τώρα είμαστε υποχρεωμένοι να δεχθούμε την διαδικασία που μας επιβάλλουν οι χώρες μέλη. Ωστόσο, θα έρθω σε ορισμένα σχόλια που έγιναν. Ο κύριος Μπούσουτιλ είπε και δικαίως ότι το δικαίωμα σιγής συμπληρώνεται τώρα από τις χώρες μέλη. Υπάρχουν όμως πολλά άλλα τα οποία λείπουν και στην αρχική οδηγία υπήρχε μια δυσαναλογία ανάμεσα στα δικαιώματα εκείνα τα οποία διαλαμβάνονται στην οδηγία, στο σύνολό τους και σε εκείνα τα οποία περιλαμβάνονται στην παραγράφο 3. Γι' αυτό το λόγο όλα τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην οδηγία τα βάζουμε στην παράγραφο 3 ώστε να μην υπάρξουν κενά. Αυτό είναι σημαντικό. Σημαντικό είναι επίσης το θέμα πώς εξηγώ τα δίκαια όταν κάποιος δεν μπορεί να διαβάσει, όταν κάποιος έχει διανοητικές ε, αδυναμίες. Το θέμα είναι επίσης, σημαντικό θέμα είναι επίσης η εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού. Πότε θα πρέπει να χορηγείται στον ύποπτο η ενημερωτική επιστολή. Θα πρέπει να γίνεται αυτό σε ένα πρώιμο στάδιο. Το θέμα της αρχής που είναι υπόχρεη να ενημερώσει μπορεί να το λύσει ίσως το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλουμε βέβαια εμείς να το ξεκαθαρίσουμε τώρα, μπαίνουμε πάλι στον χώρο της εναρμόνισης. Και τότε αρχίζουν δυσκολίες με τούτην εδώ την, με τούτην εδώ την οδηγία. Η κυρία Βίξτρομ αναφέρθηκε και σε ορισμένα θέματα που απαιτούν κάποιες γλωσσικές διευκρινήσεις. Έχουμε κάνει εμείς σχετικές προτάσεις και για, την έννοια charge και για την έννοια case, υπόθεση, που δίνεται επίσης διαφορετική έννοια σε διάφορες χώρες μέλη. Προτείναμε διαφορετικούς ορισμούς που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα. Το ζήτημα επίσης ε, της ενημέρωσης για μικρά αδικήματα, παραπτώματα κλπ. Επίσης είναι σημαντικό και αυτό γιατί και εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα σε μικρές παραβιάσεις ε, ή παραβάσεις να, υπάρχει το, να υπάρχουν τα δικαιώματα αυτά. Θα πρέπει και αυτό να διευκρινιστεί σε ορισμένες παραγράφους. Το θέμα της εναρμόνισης νομίζω ότι είναι σημαντικό να συμφωνήσουμε με, με την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τον καθορισμό δικαιωμάτων, και αυτό δεν σημαίνει καθόλου εναρμόνιση δικαιωμάτων, αν δηλαδή θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τέλος της roadmap, ώστε να περιληφθούν όλα τα δικαιώματα τα οποία μέχρι τότε θα έχουν εγκριθεί ή θα έχουν εναρμονιστεί στην ενημερωτική επιστολή ή εάν για παράδειγμα το ζήτημα της επαφής με κάποιον οικείο ε, πρέπει από τώρα να περιληφθεί, έστω και αν ρυθμίζεται διαφορετικά σε διάφορες χώρες μέλη. Θα περιμένω τις επόμενες μέρες διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Thank you. Και εν τέλος ευχαριστώ πολύ, εν τέλει συγγνώμη ευχαριστώ πολύ για τις ε, πολλές υποδείξεις. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι φτάνουμε στο τέλος αυτού του τμήματος τη συνεδρίαση της ΛΥΜΠ. Φαίνεται ότι τα καταφέρνουμε εγκαίρως. Η κυρία Σίπελ. Η κυρία Σίπελ πάλι. στην αρχή της συζητήσεως του θέματος αυτού είχε ζητήσει ο Πρόεδρος προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών μέχρι τις 12 Ιανουαρίου επειδή πρόκειται πραγματικά μόνο για την ενημέρωση, πληροφόρηση και δυστυχώς όχι για την, πληρο... για την εναρμόνιση, θα θέλαμε πραγματικά να έχουμε μια πρώτη προσανατολιστική ψηφοφορία, orientation vote, ήδη τα τέλη Ιανουαρίου, ώστε να ξέρουμε πώς θα προχωρήσουμε στον τριμερή διάλογο με τις χώρες μέλη και με την Κομισιόν. Αυτά εν Δεν θέλω να ανατρέψω το χρονοδιάγραμμα, αλλά δεν είναι κάπως πολύ σύντομη αυτή η προθεσμία. Είναι αμέσως μετά από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Για την έκθεση για τους Ρωμά είχατε 10 Ιανουαρίου. Και εσείς τώρα είπατε... Α, 12, ε, μάλιστα. Ίσως προξενήσει πρόβλημα αυτό. Δεν θέλω βέβαια να ανατρέψω το χρονοδιάγραμμα της εισηγητρίας, αλλά ας το λάβουμε υπόψη μας. Η συγκήτρια είναι ανοιχτή. Ε, αν η προθεσμία καταθέσεως τροπολογιών είναι επαρκής ή μήπως θα έπρεπε να παραταθεί επειδή, επειδή είναι ακριβώς μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων. Η κυρία Ζήπελ, εγώ θεωρώ ότι όσοι εργάζονται πάνω στην εκθέση αυτή έχουν ήδη κάνει τη δουλειά τους και πολλοί βουλευτές δεν θα πάνε και τρεις εβδομάδες διακοπές για μένα θα ήταν σημαντικό, εάν δεν υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξει να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε την ε, προθεσμία αυτή. Καλά λοιπόν, λέει ο Πρόεδρος, τότε η κατάθεση τροπολογιών ε, θα πρέπει να γίνει μέχρι τις 12 πρώτου, 12 το μεσημέρι. Προσεγγίζουμε το πέρα των εργασιών, το τελευταίο μέρος τώρα Έχουμε αναβάλει ορισμένα θέματα για την επόμενη ε, συνάντηση. Ας σας πω στα διάφορα προσδιορισμών εισηγητές. Διαβάζω απλώς. Οι αποφάσεις που ε, λήφθηκαν στις συναντήσεις των συντονιστών, στις προηγούμενες. Πρώτα, καθιέρωση ενός μηχανισμού αξιολογήσεως για την αξιολόγηση του Σέγγεν. Κοέλιο, δεύτερο πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σέγγεν στην Δημοκρατία της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, Κοέλιο. Τρίτο, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την προστασία δεδομένων. Εισηγητής, Άξελ Φως. Τέταρτο, επιθέσεις κατά πληροφοριακών συστημάτων. Εισηγητής, Μόνικα Χόλμαϊρ. Πέμπτο, κατάλογος ταξιδιωτικών εγγράφων που επιτρέπουν στον κάτοχο να διαβεί τα εξωτερικά σύνορα και που μπορεί να, σε αυτά να πρεστήθεται και βίζα, προξενική θεώρηση. Εισηγητής Τάνια Φαγιόν. Έκτο. Γιάν Μούλτερ για την ε, ε, εμπορία διαφόρων υλών. Επίσης, το επόμενο, η κυρία Φρασίκο Βαμπένοβα. Τέλο, ο, ε, γνωμοδοτήσεις τώρα, μεταναστευτικέ ροές. Ελένη Φρότρο. Δεύτερο, πρόθεση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. βιτσιούτε Τρίτο, ενιαία αγορά για Ευρωπαίους συγητής Βαντεκάμπ. Τέταρτο, ασφάλεια αερομεταφορών ιδιαίτερα σκάνερ. Η συγήτρια Σαρτζεντίνη. Τέλος, Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Η συγητής Αλεξάνδερ Άλβαρο. Αυτά για την ώρα. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 10 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες και αν δεν έχετε ε, επιφυλάξει ενστάσεις. Αυτά λοιπόν εγκρίνονται. Σας λέω στο Στρασβούργο. Ε?